Ε, συνεδρίαση αυτής θα δοθούν για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στου αποδέκτε του. Η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει διακοπεί και σας εύχομαι σε